η ερμηνεία αυτή. Μία ακόμη ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας με ενημέρωσαν για την εκλογή της κυρίας Κριστίν Ρεβό Νανών Μονεφουά που θα αντικαταστήσει τον κύριο Ντεζίρ από τις 9 Απριλίου 2014 βάσει του άρθρου 7 άρθρο 1 για την εκλογή των Ευρωβουλευτών βάσει Καθολική Άμεση ψηφοφορία και του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 4 του εσωτερικού κανονισμού το Ευρωκοινοβούλιο σημειώνει την εκλογή τη κυρία Ζεμπό από τις 9 Απριλίου 2014. Εύχομαι το καλώς ήρθατε στην ε, συνάδελφο και θυμίζω ότι βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και εφόσον οι αρμοδιότητες της δεν έχουν να εξελιχθεί ή δεν υπάρξουν αντιρρήσεις Να θα υπάρξει ένα πρόβλημα με την ανάληψη καθηκόντων. Μπορεί να ασκήσει πλήρως τι αρμοδιότητε τη, εφόσον υπογράψει τη δήλωση ότι δεν θα υπάρξει ανάληψη καθηκόντων που είναι ασύμβατα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού. Και τώρα να περάσουμε στην συζήτηση. Με πρώτο σημείο για την κοινή μας συζήτηση την Τραπεζική Ένωση. Εκθέσεις Huckmark πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση επιστοτικών ιδρυμάτων